Colleagues. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Είμαστε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Ψηφοφορία για το διορισμό του Προέδρου της ΕΣΓΑΠ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συμβουλευτικού Συμβουλίου ε, για τη διακυβέρνηση του τομέα της στατιστικής. Εχθές έγινε η ακρόαση, μετά έγινε η θετική αξιολόγηση ε, και κλεισμένο των θυρών και τώρα ολοκληρώνει τη διαδικασία με την επίσημη ψηφοφορία επί τη βάση της πρότασης του Συμβουλίου να αναλάβει την Προεδρία της ΣΓΑΠ ο κύριος Μάρτι Χετεμάκη. Θα ήθελα by... Θα ζητήσω από τους συναδέλφους να ψηφίσουν ο κυρός. Υπέρ του διορισμού του κυρίου Χετεμάκη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον κύριο Χετεμάκη. Now We can move to point Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 9. Οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων, για τη γνώμη της Επιτροπής για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της Ευρωζώνης. πιο συγκεκριμένα των 16 χωρών μελών της Ευρωζώνης και φυσικά την αναθεώρηση των κανονισμών της δέσμης των 2 μέτρων και των 6 ε, μέτρων όπως παρουσιάστηκαν και φυσικά και εν ώψη και της ε, ανακοίνωσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος Δομπρόσκης και ο Επίτροπος Μασκοβισή και μας παρουσίασαν και μας είπαν ότι θα γίνει τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι η συζήτηση που μόλις έγινε για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης μας καθορίζει πολύ σαφούς και συνεκτικούς ε, οικονομικούς ε, στόχους πολιτικής και στρατηγική. Και σε ό,τι αφορά το σχέδιο προπολογισμού, είναι σαφές ότι αποτελεί αναπόσπαστο του τμήμα της προσέγγισης αυτής. Αυτό ήδη αναφέρθηκε. Και τώρα, κ. Μουσκοβισή, θα προσπαθήσει να επισέλθει στις λεπτομέρειες και να μας πει ποια είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξέταση αυτών των αυστηρών σχεδίων στο πλαίσιο της αλλαγής για μια ουδέτερη στάση σε όλη την Ευρωζώνη, αλλά με διαφοροποιήσεις. Σίγουρα αυτό θα είναι ενδιαφέρον σημείο το οποίο και θα συζητήσουμε. Ένα άλλο μεγάλο θέμα θα είναι ασφαλώς η κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών. όπου δεν διαπιστώθηκε σοβαρή παράβαση σε κανένα κρατός μέλος, αλλά 7 κρατημέλη διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Και έχουμε και αυτό το νέο στοιχείο, ο ρόλος ε, που παίζει η δέσμευση στις διαθετικές αλλαγές. Ενδιαφέρον. Σύνδεσμος ενδεχομένω μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής πολιτικής, δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο στοιχείων. Νέα λοιπόν ενδιαφέροντα στοιχεία και θα δώσω πάρα αυτά τον λόγο στον Επιτρόπο Μοσκοβασί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Μόλις ε, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συναδέλφους Βάλτης Ντομπρόσκης και τη Μαριάν Τάισεν που μας επέτρεψε λίγο να καθορίσουμε το συνολικό πλαίσιο ε, το οποίο ε, βασίζεται στη συνοχή. Και τώρα θα ήθελα να ε, σας πω δύο λόγια για την ανταλλαγή απόψεων που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ε, για τα σχέδια των προπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Καταρχάς, θα ήθελα από πλευρά ε, μεθοδολογία να κάνω μια σαφή διάκριση μεταξύ δύο διαδικασιών που ναι μεν είναι αλληλένδετες αλλά ταυτόχρονα είναι και ανεξάρτητες. Καταρχά πρέπει να προετοιμάσουμε το επόμενο έτος. Είναι η διαδικασία που προκύπτει από τη δέσμη των δύο μέτρων που θέλει να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα σχέδια προπολογισμού των κρατών μελών και αυτό γίνεται με την αξιολόγηση των σχεδίων προπολογισμών για το 2015 ε, και υπενθυμίζω όπω είπε και ο πρόεδρο, ότι κάποια προγράμματα προπολογισμών δεν απορρίπτουν είχαν τα τέλη Οκτωβρίου λόγω ε, πολύ σοβαρής ε, από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι σέβονται απολύτω το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Απλώ είμαστε σε ένα άλλο στάδιο αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Αυτό βέβαια είναι πάντα πιο περίπλοκο και εξαρτάται και από την κατάσταση των κρατών μελών. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι δράσει οι οποίε έγιναν για το 2014 στα πλαίσια τη διαδικασία υπερβιλικού ελλείμματο και αυτό το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε ε, ε, είναι να το εξετάζουμε μέχρι τα μετά ο Μάρτιο του 2015. Τώρα, να περάσω στην ουσία ποιε είναι οι συνέπειε για τι διαδικασίε του υπερβολικού ελλείμματο, οι οποίε πρέπει να συζητηθούν ε, μόλι έρθει κατάλληλη στιγμή. Για τρει χώρε, για τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει στι αρχέ Μαρτίου του 2015 την κατάστασή του σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Και αυτό θα γίνει με βάση αρκετών στοιχείων, καταρχά την εκτέλεση του προπολογισμού του 2014, για να δούμε κατά πόσον εφαρμόστηκαν ε, συγκεκριμένε δράσει στι οποίε σα αναφέρω, μετά την ολοκλήρωση των δημοσιονομικών κανονισμών για το 2015 για να δούμε εάν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για το 2015 παρκούν και επίσης θα δούμε και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσαν οι αρχές στις επιστολές που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δημοσιοποιήθηκαν και είναι διαθέσιμες φυσικά ε, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις μας. Αυτά τα τρία κρατημέλη, να σας υπενθυμίσω ότι δεσμεύτηκαν στο πιο υψηλό επίπεδο μέσω των πρωθυπουργών τους να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης στις αρχές του 2015, οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνέπειες και για την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αλλά φυσικά και στην ανάπτυξη. Από πλευράς μας, και αυτό φυσικά θα το συζητήσουμε, αυτή η διαδικασία εγγυάται και την συνέπεια και την ε, ε, αξιοπιστία των κανόνων μας. Αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες ε, στα κράτη-μέλη και αφετέρου δεν έχουμε και δεν θελήσαμε άλλωστε να λάβουμε βεβαιασμένες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να αμφισβητηθούν αυτή τη στιγμή γίνουν γνωστά τα οριστικά στοιχεία. Αυτά κυρίως όσον αφορά το 2014 για τα οποία δεν έχουμε ακόμα εξορισμού πλήρη στοιχεία. Η Επιτροπή ε, δίνει σε, στα 16 κράτη-μέλη της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωζώνης την άποψή της για τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2015 πριν ε, την οριστική έγκρισή τους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα αποτέλεσμα της ανάλυσης, της ανάλυσης μας είναι σαφή. Θα πρέπει να, καταρχάς να ομαδοποιήσουμε. Έχουμε πέντε χώρες οι οποίες τηρούν απολύτως το σύμφωνο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι κάτω χώρες και η Σλοβακία. Στην περίπτωση της Γερμανίας, και αυτό σχετίζεται και με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως ε, για το μηχανισμό επαγρύπνησης και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, διαπιστώνουμε ότι ε, υπάρχει σημαντικό ε, περιθώριο στον προπολογισμό και οι ανάγκες για επενδύσεις και κυρίως τα επιτόκια θα επιτρέπουν να υπάρχουν αύξηση των επενδύσεων. Τέσσερις χώρες, η Εστονία, η Λετωνία, η Σλοβενία και η Φιλανδία παρουσίασαν σχέδια προπολογισμού τα οποία γενικώ θεωρούμε ότι συμμορφούνται. Διαπιστώνουμε όμως ότι 7 χώρες, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Πορτογαλία, ε, έχουν ένα σχέδιο προπολογισμού που ελοχεύει ο κίνδυνο μη συμμόρφωση. Το σχέδιο προπολογισμού τη Ισπανία, τη Γαλλία και τη Πορτογαλία δημιουργεί κινδύνου ε, κυρίω όσον αφορά των απαιτήσεων τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο που εφαρμόζονται στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα για τη Γαλλία, οι πληροφορίε που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υποδηλώνουν ότι η Γαλλία θα μπο... ίσως δεν έχει λάβει κάποια μέτρα λόγω των φαινομένων του 2014 και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην συμμορφούνται με τους κανόνες και τις απαιτήσει ε, της ε, διόρθωσης που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει και πολύ συγκεκριμένη επιτήρηση. Το Βέλγιο και η Ιταλία βρίσκονται σε μια διαφορετική κατάσταση διότι ε, βρίσκονται στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου, ελοχεύει ο κίνδυνος να μην συμφωνούν ε, να σεβαστούν τον άλλο κανόνα του δημοσίου χρέους, ένας κανόνας ο οποίος είναι πάρα πολύ απαιτητικός δεδομένης κατάστασης στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Έχουμε ισχνή ανάπτυξη και πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Καλούμε λοιπόν τις αρχές των 11 χωρών να λάβουν στα πλαίσια των διαδικασιών των εθνικών τους προπολογισμών μέτρα προκειμένου να ε, διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ε, συμμόρφωση στον προπολογισμό του 2015 με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πέραν ε, από τις γνώμες για το σχέδιο προπολογισμού, παρουσιάζουμε επίσης και ανάλυση της κατάστασης και προοπτικές για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης συνολικά. Και επίσης και κάποια συνολικά στοιχεία για το τους προσανατολισμούς ε, ε, για τον συνολικό προϋπολογισμό και αυτή η διαδικασία θέλει να ενισχύσει την διάσταση της Ευρωζώνης ε, και τα θέματα της επιτήρησης του προπολογισμού. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτή τη στιγμή. Τα σχέδια προπολογισμού δείχνουν μία μείωση λοιπόν στο συνολικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης ε, μετά από τη μείωση σε κάτω από το 3% του ΑΕΠ ε, το 2014 το συνολικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη ε, θα μειωθεί κατά 2,6% το 2014 και 2,2% το 2015. Το συνολικό ποσοστό χρέους του 2015 προγραμματίζεται, αναμένεται να παραμείνει το ίδιο ε, με την τιμή που εκτιμούμε για το τρέχον έτος, 92,5% του ΑΕΠ. Και χάρη στις ε, προσπάθειες μας στο παρελθόν, και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι έχουμε πλέον μια ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική. Και φαίνεται ότι αυτό είναι το πλέον κατάλληλο. Και αυτό μας βοηθά να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων βιωσιμότητας, δεδομένου του υψηλού ποσοστού χρέους και, ε, και ανησυχίες κυκλικής σταθεροποίησης λόγω της χαμηλής ανάπτυξης, του χαμηλού πληθωρισμού και φυσικά και των περιορισμών που ε, προκύπτουν από την νομισματική πολιτική. Ωστόσο, η αξιολόγηση των σχεδίων επιβεβαιώνει ότι αρκετά κράτη-μέλη αναμένεται να μην τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ κάποιες άλλες αναμένεται να επιτύχουν υπερβολικά τους στόχους αυτούς. Και αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη συνολική ε, ουδέτερη δημοσιονομική στάση στην Ευρωζώνη, όπου κάποια κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εκμετάλλευση του δημοσιονομικού περιθωρίου κάπου αλλού, ε, θα χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση, συνεπώς, επισημαίνει πάρα πολύ ε, σημαντικά την ανάγκη για συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και για το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη που παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου. Αυτά για τις γνωμοδοτήσεις, και, για τις γνώμες μας και για τη συνολική κατάσταση. Και τώρα να σας πω δύο λόγια για κάτι ακόμα που συζητάει η Επιτροπή σα, η επισκόπηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωσή της για την αξιολόγηση της εφαρμογής της δέσμης των 6 και των 2 μέτρων, ε, τη λεγόμενη επισκόπηση της οικονομικής διακυβέρνησης και η οικονομική και η ε, χρηματοπιστωτική κρίση ε, αποκάλυψαν πολύ σημαντικές αδυναμίες στην αρχική ε, δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως επισημάνει και η κυρία Μπερές ε, στο έγγραφο εργασίας για την, ε, για την επισκόπηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Λήφθησαν κάποια μέτρα για, με βάση τα όσα θεωρήθηκαν ότι ήταν εφικτά πριν από κάποια χρόνια. Η Ευρωζώνη πιέστηκε από τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού του ESM για να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα, τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε την χρηματοπιστωτική, το χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό και την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης για να ενισχύσουμε την οικονομική ε, διάσταση και το συντονισμό σε θέματα προπολογισμού. Τώρα, οι δέσμοι των 6 και των 2 μέτρων οδήγησαν στην ενίσχυση τη ε, δημοσιονομική εποπτείας με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, ε, καθώ επίση και αντιμετώπιση των προβλημάτων κάποιων χωρών που αντιμετώπιζαν προβλήματα με την δημοσιονομική σταθερότητα. Με βάση τις νομικές απαιτήσει στα διάφορα νομοθετήματα έγινε επισκόπηση των νέων αυτών μέσων. Ε, η ρήτρα αναθεώρηση απαιτεί αξιολόγηση τριών στοιχείων. Την αποτελεσματικότητα των κανονισμών, δεύτερον, σε ποιο βαθμό οι κανόνε συνεισέφεραν στην πρόοδο σε στενό συντονισμό με τις οικονομικές πολιτικές και τρίτον, σε ποιο βαθμό οι κανόνες συνεισέφεραν και στη βιώσιμη οικονομική σύγκληση. Λόγω του περιορισμένου ε, χρόνου, λόγω μετά τη θέση σε ισχύ, η εμπειρία μας με την εφαρμογή του νέου οικονομικού συστήματος διακυβέρνησης είναι αρκετά περιορισμένη και κάποια συγκεκριμένα εργαλεία όπως για παράδειγμα η διαδικασία υπερβολικού, ε, υπερβολικών ανισορροπιών δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί. Το σύστημα μέχρι το ουδέ έχει εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες ε, κατά τη διάρκεια ή μετά από μια πολύ σοβαρή κρίση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η επισκόπηση πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι αρκετά σύντομη, ε, αφορά συγκεκριμένα στοιχεία, εξετάζει το παρελθόν και επικεντρώνεται και στην εφαρμογή των νέων μέσων. Συζητά ξεχωριστά τα θέματα της δημοσιονομικής εποπτείας, των μακροοικονομικών ανισορροπιών και το πλαίσιο για τις χώρες οι οποίες βιώνουν πολύ σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τη δημοσιονομική του σταθερότητα. Η αναθεώρηση η επισκόπηση μάλλον επισημαίνει και τις ε, βελτιώσεις που εισήχθησαν από τα δέσμη των έξι και των 2 μέτρων, έχει εμβαθύνει ε, την οικονομική διακυβέρνηση και έχει συνεισφέρει στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τη ε, δημοσιονομική εξυγίανση και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ισορροπιών. Όπω ε, έπηξε επίση και από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή ΕΚΟΝ εδώ στι 4 Νοεμβρίου, υπάρχει σαφώ περιθώριο βελτίωση. Αυτό σχετίζεται με την περιπλοκότητα του συστήματο, ε, κάποια εργαλεία έχουν αλληλοεπικαλύψεις και την περιπλοκότητα των συγκεκριμένων εργαλείων συγκεκριμένα, Όπω για παράδειγμα το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Η περιπλοκότητα μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στη διαφάνεια και στην εφαρμογή. Η επισκόπηση επίση αναφέρεται στην ανάγκη να διασφαλίσουμε ιδιοκτησία και τις ε, ε, προσπάθειες από πλευράς πολιτικής στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων ε, βάσει ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της μεσοπρόθεσμης του MIP. Και επίσης πρέπει να υπάρχει καλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κοινοβουλίων για να έχουμε μεγαλύτερη νομιμοποίηση το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πλήρες δυνατότητές τους μόνο εάν υπάρχει ε, διοκτησία όλων των ενδιαφερομένων μερών και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι το βασικό θεσμικό όργανο που μπορεί να διασφαλίσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο λήψης αποφάσεων σε οικονομικά θέματα και θα ολοκληρώσω με αυτό διότι μακρηγόρησα λίγο. Θεωρούμε ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί την αρχή του διαλόγου και τη συζήτηση για την κατάλληλη άγουσα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στου επόμενους μήνες. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα και με τους συζητητές και τους κοιόδη συζητητέ για τα θέματα αυτά και θα ήθελα να ε, πω σε όλους ότι είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να συζητήσουμε μαζί σας, ε, θέλουμε να ακούμε τις απόψεις σας και θέλουμε ε, να δούμε και τι μπορείτε να συνεισφέρεστε, διότι αυτή είναι μια διτή προσέγγιση. Καταρχά υπάρχει αυτή η έκθεση, η οποία θα μπορούσε ίσω να πούμε ότι είναι περιορισμένη και είναι απλώ βασισμένη σε στοιχεία και από εκεί και πέρα ε, το μακρόπνο όραμα ε, και ο πρόεδρο Γιούνκερ είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σε αυτό. Σα ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στον πρωτομιλητή. Έχουμε πέντε λεπτά κάθε φορά για το γύρο ερωτήσεων και πέντε ε, λεπτά για τι απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επιτροπέ, ο κύριος Φερμπέρ. Ανακύπτουν κάποιες ερωτήσεις στο μυαλό μου. Θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το six pack και το ΤΟΥΠΑΚ. pack Προβλέψαμε σαφείς ε, προθεσμίες για μια διαδικασία κατά τη βούληση των κρατών μελών που μια διαδικασία που προβλέπει αυτοματισμό. Και αυτό γιατί εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφυλάκα των συνθήκων προκειμένου να φροντίσει την ε, τήρηση, για την τήρηση των κανόνων. Γιατί από το παλιό Σύμφωνο θεραότητας και Ανάπτυξης είδαμε ότι τα κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα να ερμηνεύουν τους κανόνες και αν υπήρχε πολιτική ανάγκη αποφάσεων ήταν ε, θέμα του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών να αποφασίσει κατά του αυτοματισμού αυτού. Τώρα λοιπόν βλέπω ότι το Μάρτιο θα γίνει η διαδικασία για τον δημοσιονομικό έλεγχο. Ε, λοιπόν και θα ήθελα να έχω συγκεκριμένη απάντηση. Γιατί οι κανόνες στο συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποδυναμώνονται. Αυτή έπρεπε να φροντίσει να τηρούνται οι κανόνες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια να μην φροντίζει για την τήρηση των κανόνων. Δεύτερη ερώτηση. Είχαμε ενίσχυση του προληπτικού σκέλους. Αυτό είχε προβλεφθεί. Προκειμένου να μην καταλήξουμε σε προβληματικές καταστάσεις. Και τώρα έχω κάπως την, αίτηση, την αίσθηση στις ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις και στις συζητήσεις για τη μεταξέλιξη του 2-pack και του 6-pack ότι και αυτό συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο αποδυνάμωσης. Τι να το κάνουμε το ισχυρό προληπτικό σκέλος αν δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή. Διευκρινίστε μας λοιπόν σας παρακαλώ τι γίνεται με τις ε, συνθήκες πλαίσιο 2014 σε ό,τι αφορά την αποδυνάμωση των κανόνων αυτών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Euh, Οι ερωτήσεις του κ. Φέρμπερ είναι μάλλον ε, από ό,τι υποπτεύομαι πολύ πιο συγκεκριμένε από όπως τις παρουσίασε. Θα απαντήσω λίγο πιο γενικά. Να πω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τις απόψεις της, έχει τις γνώμες της ε, και θεωρεί ότι πραγματικά είναι ο θεματοφύλακας των κανόνων. Και αυτό ακριβώ μα οδήγησε και στι αποφάσει που λάβαμε με τον κύριο Και αυτό πάντα θα γίνεται, σα διαβεβαιώ για κάποιες χώρες ε, διαπιστώσαμε ότι ακόμα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε άποψη ε, για να αποφύγουμε και τυχόν ε, λάθη. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ε, κάποιο περιθώριο για τρεις χώρες στις οποίες αναφέρθηκα και στις οποίες μάλλον ε, αναφερθήκατε κι εσείς. Ε, έχουμε μέχρι το Μάρτιο του 2015 περιθώριο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ακόμα κι αν υπάρχει αυτός ο επιπλέον χρόνος, ε, μια καθυστέρηση, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί χαμένος χρόνος, διότι θα το χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω κράτη-μέλη για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με δημιουργικό τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες ε, και θέλει να δει αν υπάρχουν διορθωτικά μέτρα τα οποία λήφθησαν στο παρελθόν, αν υπάρχουν συγκεκριμένε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για το μέλλον και αν είναι αρκετά δημιουργικές και οδηγούν ανάπτυξη και φυσικά εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Και βεβαίως υπάρχει και ένα συγκεκριμένο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, ε, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε καθήκοντα από 1η Νοεμβρίου, το οποίο ίσως έχει περιπλέξει λίγο τη διαδικασία ε, της αναδρομικής διαδικασίας ε, για το 2014. Ε, με το Βάλτις Δομπρόσκης αυτό που κάναμε ήταν να, να αποφασίσουμε ήδη ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα την επόμενη χρονιά. Είναι πολύ πιο εύκολο να διορθώσει κάποιο ένα προπολογισμό και αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι επίκριση κατά τη προηγούμενη επιτροπή αν ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο από ότι αν ξεκινήσουμε το Νοέμβριο. Γι' αυτό ακριβώ και ε, υπάρχει αυτή η επιπλέον προθεσμία. Ε, τηρούμε του κανόνε μα, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε παραβίαση των κανόνε, γίνεται σεβαστοί κανόνε και και με αυτό το πνεύμα θα λαμβάνουμε αποφάσεις με όλο το οπλοστάσιο στη διάθεσή μας δεν αποκλείουμε κανένα όπλο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής η Ελίζα Φεραίρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Δύο ερωτήσει έχω να σας θέσω. Η πρώτη. Η Επιτροπή από πλευράς μου δεν θεωρώ ότι εφαρμόζει την νομοθεσία όπως υφίσταται. Στο κανονισμό 1175 προβλέπονται και το σκέλος, το, ρυθμιστικό, το προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του συμφώνου. Έχουμε και ρήτρες διαφυγής. Και στα δύο σκέλη για περιπτώσεις εξαιρετικών οικονομικών συνθήκων. Στον κανονισμό που μόλις σας ανέφερα, προβλέπονται τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούν να υπάρξουν παρεκκλήσεις από τον μεσοπρόθεσμο στόχο. Ασυνήθιστα περιστατικά, σημαντικές οικονομικές ε, δυσκολίες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και το άρθρο 5 του κανονισμού προβλέπει ότι το σύνολο των επενδύσεων θα περιλαμβάνει τον τόκο των επενδύσεων, ε, επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Ένωση και αλλαγές ε, στις ε, δαπάνες επενδύσεων. Τίποτα από αυτά δεν εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερη και δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση και θεωρώ ότι ακόμα και η επιστολή του Όλι Ρεν επιβάλλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη χρήση των ε, μέτρων αυτών που προβλέπονται από το νομικό κείμενο. Ζούμε λοιπόν θεωρώ σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει το νόμο. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, προτίθεστε να αλλάξετε την κατάσταση αυτή. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις. Επιβάλλουμε κυρώσεις στα κρατημέλη για προβλέψεις που δεν ακολουθούνται. Ή, εν πάση περιπτώσει, συζητάμε την δυνατότητα και την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων. Και κοιτώντας τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Ιρλανδία, για παράδειγμα, η ανάπτυξη για το 2014, την άνοιξη ήταν 1,3. Το φθινόπωρο 2,2 στη Λιθουανία και αναφέρω διάφορα κράτη-μέλη, πρόβλεψη ανάπτυξης για το ίδιο έτος, την άνοιξη 3,1, 2,5 την Συνόπορο, για το Λουξεμβούργο, για το 2015, 1,3 την άνοιξη, 2,2 το φθινόπωρο. Κοιτώντας την εκτίμηση του ελλείμματος, το έλλειμμα μεταξύ το κοινό μεταξύ των ε, το πληρωμών και των αναλύσεων και των ε, διαφορών είναι για την Ισπανία 1,6, 0,8 για τη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις εκτιμήσεις. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό σύστημα κυρώσεων και συστάσεων όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στις εκτιμήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Καταρχάς, ε, για την πρώτη σας παρατήρηση, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω μαζί σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ε, για να κάνει δημιουργική ερμηνεία των κανόνων, ούτε να τους ε, παραβλέπει. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να τους σεβόμαστε. Αναφερθήκατε στην ευελιξία στα πλαίσια των υφιστάμενων κανόνων να σας ε, επαναλάβω ότι θα υπάρξει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον κύριο Ντομπρόφσκης και από μένα και ε, λαμβάνουμε υπόψη και την περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων. Έχει γίνει συζήτηση από αυτόν, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένε δυνατότητες και από πλευράς διορθωτικών μέτρων αλλά και από πλευράς πρόληψης ε, κάποιων φαινομένων και υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί κάποια ευελιξία, αλλά δεν εκτιμούμε ότι σε επίπεδο της Ευρωζώνης ότι βρισκόμαστε σε κάποια έκτακτη κατάσταση η οποία θα απαιτεί, για παράδειγμα, να ε, μην έχουμε γνώμη για τις επόμενες χρονιές και να δούμε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Ίσα ίσα θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση αναχώρα που θεωρούμε ότι συνάδει και συμμορφούται με το γράμμα των κανόνων μας. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψει κάποια έκτακτη περίπτωση. Ε, υπάρχουν αξιολογήσεις, οι προβλέψεις και συνειδητοποιώ απολύτω ότι ε, έχουν υπάρξει και λάθη στο παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς και όταν παρουσιάσαμε τις προβλέψεις για την επόμενη χρονιά, ε, μαζί με τον Γιούρκη Κατάινεν, ε, ήμασταν ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε τις πολύ σημαντικές διαφορές ε, και ε, την αισιοδοξία να γίνει απεσιοδοξία την, ε, εν μία νυχτή. Προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ ιδιαίτερα. Και ο Γιώργη Κατάινεν συμφωνεί ότι οι προβλέψεις δεν θα πρέπει πλέον να παρουσιάζονται από τους επιτρόπους αλλά από τους γενικούς διευθυντές που είναι αρμόδιοι για τη χώρα κάθε φορά. Σας ευχαριστώ από το ECR. Ο κύριος Λούκε έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με ανησυχία διαπιστώνω ότι συνεχώς τονίζετε την ευελιξία των κανόνων και την επιθυμία να εφαρμοστούν με ευελιξία οι κανόνες. Λάθος αντίδραση εκτιμώ. Θα πρέπει να εφαρμόζονται πιο αυστηρά οι κανόνες. Και ο λόγος είναι ο εξής. Οι κανόνες καταρτίστηκαν σε μια κατάσταση κανονικής ανάπτυξης, φυσιολογικής ανάπτυξης, φυσιολογικού ποσοστού πληθωρισμού 2%. Είχαμε ορίσει λοιπόν το 3% ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και αυτό γιατί ξέραμε ότι η ανάπτυξη κάθε χρόνο μειώνεται 2% περίπου, λόγω πληθωρισμού. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, διαπιστώσαμε μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά και αύξηση κατά όριο 3% είχαν ορίσει οι κανόνες. Τώρα όμως δεν υπάρχει ουσιαστικά πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη. Δηλαδή το χρέος δεν μειώνεται με την νέα ε, πληθωρισμό και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες για τη νέα χρέωση. Στην έκθεση λοιπόν διαπιστώνεται ότι στην Ευρωζώνη οι νέε χρεώσει με μέσα 4,1% το 2011 μειώθηκαν σε 2,6% το έτος 2014. Αλλά αυτό το πουλάτε σαν νίκη. Στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται είναι το γεγονός ότι μέσω του πληθωρισμού δεν μειώνεται πλέον το χρέος και έτσι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί στην πραγματικότητα. Πραγματικά έχουμε αύξηση του χρέους όπως και το 2011 άλλωστε. Και αν δεν κοιτάξουμε τι γίνεται στο μέσο όρο, κοιτώντας τις χώρες όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, όπως και χώρες της Γαλλίας, όπου υπάρχει έλλειμμα μεγαλύτερο 4% του προπολογισμού και του τράχοντος έτους και του επόμενου έτους και του μεθεπόμενου έτους. Αυτό καταδεικνύει πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση. Τοποθετηθείτε λοιπόν, μήπως θα ήταν ε, απαραίτητο όχι να είμαστε πιο ευέλικτοι, αλλά και πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Ε, um, Πρώτα Πρώτα θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ποια είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε την συμμόρφωση με τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Εκτιμούμε λοιπόν ποια είναι ε, η συμμόρφωση με το Σύμφωνο Ανάπτυξης και σταθερότητα και με τι συστάσεις. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου, εκτιμούμε κατά πόσον το σχέδιο προπολογισμού εξασφαλίζει το σεβασμό των ελλημάτων που προβλέπονται από τις συνθήκη 3% και 60% σε ό,τι αφορά τη χρέωση. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει σωστή μείωση. Και κατά πόσον ο προπολογισμό συνάδει με τους μεσοπρόθεσμους στόχους, όπως ε, συστάθηκε στις αρχές του έτους από το Συμβούλιο για τα κρατημέλη στο προληπτικό σκέλος. Με μεγάλα υπερβολικά ε, ελλείμματα είδαμε κατά πόσον το σχέδιο προπολογισμού εγγυάται συμμόρφωση για τη διόρθωση του, του υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό περιλαμβάνει η εκτίμηση της προάδου και κατά πόσον όντως έχει ληφθεί επαρκής ε, ενέργειες για την ε, ανάλυση των ε, μέτρων εν λόγω. Αυτά λοιπόν έχουν ήδη ποσοτοκοποιηθεί με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το MCA και το EMC. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω δηλαδή κύριε Λουκέ είναι ότι εμείς δεν είμαστε υπέρμαχοι μιας ευελιξίας ε, ε χωρίς όρια. Ε, και δεν λέω ότι έχει ξεκινήσει από λανθασμένη διαδικασία ή από καλή διαδικασία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς εφαρμόζουμε τις κανόνες και όταν αναφερόμαστε σε ευελιξία, δεν αναφερόμαστε σε νέα ευελιξία με τον κύριο Ντομπρόσκη αναφερόμαστε σε μια ανακοίνωση η οποία ε, ακριβώς αυτό θα κάνει και αυτό είναι καλό και για τη διαφάνεια στη συζήτησή μας, είναι ευελιξία η οποία μας επιτρέπεται από τους κανόνες και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το έχω πει και εδώ σε άλλο πλαίσιο λέω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της δημιουργικής ερμηνείας των κανόνων. Δεν είμαι υπέρ ε, της ε, καταστροφής του συμφώνου. Θεωρώ ότι το σύμφωνο πρέπει να εφαρμόζεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτός είναι. Ε, έχουμε ευφυείς κανόνες και οι ευφυείς κανόνες ε, προϋποθέτουν ότι λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση στα κράτη-μέλη, ε, λαμβάνουμε υπόψη τις προσπάθειες που γίνονται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όπως είπε και η Ελίζα Φεριέρα, στην αντίθετη περίπτωση ε, τότε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα είτε για την τάδε για τη δίνα χώρα είτε για το σύνολο της Ευρωζώνης. Και να σας πω ότι το ερώτημα των επενδύσεων ετέθη και στα θέματα της παρουσίασης του ε, σχεδίου επενδύσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ που ξέρετε ότι εκεί ε, παρουσιάστηκαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ. Επίτροπε δεν απαντήσατε καθόλου, καθόλου την ερώτησή μου. Δεν την απαντήσατε. Ούτε καν αναφέρατε τον όρο πληθωρισμός. Νομίζω αντιθέτως ότι σας απάντησα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτήσατε. Ζητήσατε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ε, για να ε, κάνει ευελιξία ή για να σέβεται τους κανόνες. Ο συνάδελφος Λούκη ανησυχεί για το χαμηλό πληθωρισμό. Θα το θέσουμε στον πρόεδρο Ντράγκη αυτό. Η κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση ως πρώην εισηγήτρια του κειμένου για τις κυρώσεις και ε, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσκολία που έχετε κατά την εκτέλεση των καθιστών κόντων σας. Ποια είναι η νομική βάση για την απόφαση Απλώς και μόνον ποια είναι η νομική βάση για να καθυστερήσετε την απόφαση στο Μάρτιο για την Γαλλία. Λέτε ότι δεν θα πρέπει να είναι χαμένος χρόνος. Ναι, μεν, αλλά εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο εξέτασα τι έλεγε ο Φράνσις Μέρ το 2003 Υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας και ζητούσε χρόνο. Και είδα ότι στην απόφασή σας ότι η Γαλλία ε, βρίσκεται στη διαδικασία υπουργικού ελλείμματος από το 2009. Πραγματικά, θεωρείτε ότι είναι θέμα χρόνου και πώς μπορείτε να αιτιολογήσετε ότι ε, δεν ε, ε, ελοχεύει ο κίνδυνος να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα, διότι όταν δίνεται μια παράταση σε μια χώρα που εδώ και χρόνια δεν καταφέρνει να συμμορφωθεί προς τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Επίσης, θεωρείτε ότι μετατρέπεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ένα κοινοτικό σύστημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες συγκεκριμένε εξουσίες. Ο Μάρκους Φέρμπρερ ανακοίνωσε, επανέλαβε πολύ σωστά ότι τις αυξήσαμε. Έχουμε ένα σύστημα κανόνων και δικαιωμάτων. Όχι ένα σύστημα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχωρέστε με, εκφράζει με πολύ καλή διάθεση και είμαι βέβαιος ότι οι υπάλληλοι εργάστηκαν πάρα πολύ καλά και κανένας δεν έχει τίποτα να τους προσάψει, αλλά τελικά οι αποφάσεις σας ουσιαστικά ε, έχουν την ίδια αξία με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την ε, ε, διατήρηση της ειρήνης. Κυρία Γκουλάρ, αν κατάλαβα καλά, αν εσείς ήσασταν στη θέση μου, γιατί αυτό κατάλαβα, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι αποφάσεις μας έχουν ληφθεί από κοινού και με βάση και την έγκριση που μας έδωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ, τις είχαμε υποβάλει και κανένας ε, δεν υποχρέωνε το σώμα των επιτρόπων, ε, το άρθρο 6 νομίζω μας δίνει αυτή την εξουσία, ε, στον κύριο Ντομπρόφσκι και σε μένα. Εσείς θα είχατε πάρει τελείως διαφορετική απάντηση. Κύριε Επίτροπε, δεν σας κατηγορώ προσωπικά, το σώμα των επιτρόπων αποφασίζει. Κυρία Κουλέρ δεν αποφασίζει το Σώμα των Επιτρόπων. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και εγώ αποφασίζουμε για το θέμα αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο και ενημερώθηκε με το Σώμα των Επιτρόπων και ο Πρόεδρος των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε στη διαδικασία λήψης απόφασης. Είναι μια κοινή απόφαση μετά από μια εις βάθος συζήτηση. Εσείς θα είχατε λάβει άλλη απόφαση ίσως. Εγώ σας εξηγώ γιατί λάβαμε τη συγκεκριμένη και σας την εξηγώ η ε, απόφαση παράτασης ε, προέκυψε από εμά. Δεν είμαστε οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είμαστε θεματοφύλακα των συνθήκων και πρέπει να εφαρμόσουμε τις συνθήκες. Για να αποφασίσουμε για κυρώσεις ή για να αποφασίσουμε να μην υπάρχουν κυρώσει, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι, επαναλαμβάνω βέβαιοι, ότι για το 2014, και αυτό είναι, πρόκειται για το άρθρο 126, 8 και 9 ε, του κανονισμού, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει βεβαιότης ότι δεν υπήρξαν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα το 2014. Η αίσθησή μας, και αυτό το λέω εδώ και διευκρινίζεται και στη γνώμη μας, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι τα μέτρα ελήφθησαν, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι. Και σκεφτείτε το εξής μετά από πολύ περίπλοκους υπολογισμούς υπάρχουν μέθοδοι ε, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Και διαπιστώνουμε ότι την δεδομένη χρονική στιγμή ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος μας ανησυχεί πάρα πολύ, οι πολύ ισχνές επενδύσεις ε, και τα μέτρα όλα αυτά λοιπόν έχουν ληφθεί. Ποια είναι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλει κυρώσεις πριν να γνωρίζουμε τα οριστικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν το οποίο αποτέλει το κίνητρο για την απόφασή μας και να δώσουμε αυτή την παράταση των τριών μηνών είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα οριστικά στοιχεία επί του ζητήματος. Το επαναλαμβάνω εδώ επειδή εμεί δεν είμαστε τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό ο χρόνο δεν θα είναι χαμένο χρόνο ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε σε αυτή τη συμπερίπτωση για τη χώρα την οποία αναφέρεται και από την οποία καταγόμαστε και οι δύο. Εάν λοιπόν προκύψει ότι δεν ληφθούν μέτρα για το 2014 και το επαληθεύσουμε αυτό ότι ε, και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για το 2015 δεν επαρκούν και ότι ε, οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα δεν επαρκούν, τότε ε, στη δεδομένη χρονική στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Μαρτίου θα αναλάβει τις ευθύνες της και ε, εάν χρειαστεί θα επιβάλλει και κυρώσεις. Θεωρούμε ότι αυτά τα οποία αποφασίσαμε συνάδουν με τους κανόνες ε, και θα είμαστε ακόμα πιο αυστηροί σε περίπτωση που δεν όπου επαληθευτούν αυτά από τα οριστικά στοιχεία. Ε, υπάρχει λοιπόν η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και υπάρχει και μια πεποίθησή μου, την οποία έχω επαναλάβει και άλλες φορές. Το πνεύμα των κανόνων μας δεν είναι να είναι κανόνας οι κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι σε περίπτωση... Ε, ε, αποτυχίας. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που και πάλι δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη, επαναλαμβάνω, ε, είναι να ε, προσαρμόζονται τα κράτη-μέλη. Και εάν υπάρχουν προβλήματα, για τα οποία δεν είμαστε ακόμα πεπισμένοι, υπάρχουν κυρώσει και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και αν πρέπει να εφαρμοστούν, θα υπάρχουν κυρώσει. Αλλά, αν μπορέσουμε να τα αποφύγουμε, ακόμα καλύτερα. Και ο επικοδομητικό διάλογο σίγουρα είναι καλύτερο. Κύριε Επίτροπε, εγώ ήμουν η εισηγήτρια για τις κυρώσεις, δεν θα με εξηγήσετε εσείς το κείμενο. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι γιατί χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να εκτιμήσετε τα οριστικά στοιχεία της Γαλλίας και της Ιταλίας και θεωρείτε ότι για τις άλλες χώρες έχετε οριστικά στοιχεία. Δεν έχετε ούτε για τις άλλες χώρες, επομένως θα πρέπει να σταματήσει ο χρόνος για όλες τις χώρες μέλη την ίδια στιγμή. Για τις άλλες χώρες δεν υπάρχουν προβλήματα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι παρκώς σαφή, για την περίπτωση της Γαλλίας δεν είναι. Επομένως, θεωρήσαμε, και εσείς, ούτε εσείς τα έχετε τα οριστικά στοιχεία για το 2014, δεν τα έχει κανείς. Επομένως, θα πάρουμε αποφάσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν όλα αυτά είχαν εξεκηγήσει νωρίτερα, εάν είχαν ευαισθητοποιεί χώρες μέλη στην υπόθεση αυτή των μέτρων, το συζήτησα και με τον κύριο Κατάινεν, δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση και ξέρω πώς γίνεται ο διάλογος με τα διάφορα κράτη-μέλη και ξέρω και τους Γάλλους και τους Ιταλούς πολύ καλά πώς έγινε ο διάλογος. Ο κύριος Βιέγκας, εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστεράς. Ε, Εμείς δεν συμφωνούμε με το Σύμφωνο Σταθερότητας και όλη τη διακυβέρνηση ως διαδικασία. Ιδιαίτερα αυτό είναι ένας, ένας περιοριστικός αυτός ε, δυνάμεων που δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντά μας. Είναι ένα πλήγμα κιόλας ε, κατά της ε, κρατικής κυριαρχίας και το, του δικαιώματος να αποφασίζουμε για το μέλλον μας αντιδημοκρατικός ο χαρακτήρας αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκαλύπτει μια κατανομή ασύμετρη της εξουσίας ε, μεταξύ των κρατών μελών. 2003-2004 όταν καθορίστηκαν οι κανόνες για το έλλειμμα από την Γερμανία και τη Γαλλία καταργήθηκε το σύμφωνο όταν βρισκόντουσαν άλλες χώρες υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Τα τελευταία ε, χρόνια 24 κράτη-μέλη αντιμετώπισαν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο ευρώ, ζώνης ευρώ, 11 χώρες από τις 16 δεν υλοποιούν τους κανόνες και κανονισμούς. Και εδώ πρέπει να ερωτήσουμε, τι δεν πάει καλά, οι κανόνες, όλες οι χώρες μήπως φταίνε που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτούς τους ίδιους κανόνες και βρίσκονται στο περιθώριο της νομιμότητας. Και πραγματικά εμείς είναι η αρχή επί της οποίας δεν συμφωνούμε. Δηλαδή τα εγχειρίδια της ε, νεοφιλελεύθερης οικονομίας που αναγκάζουν τα κράτη να περιορίζονται, να συρρυκνώνονται με αυτόν τον τρόπο και να, εκπονούν, να μην μπορούν να εκπονήσουν τις δικές τους στρατηγικές ανάπτυξης. Και σύμφωνα με τις εκθέσεις που αναλύουμε εδώ, και το σημειώνω εγώ αυτό, οι χώρες της ζώνης ευρώ αυξάνονται λιγότερο σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται εκτός ζώνης ευρώ και έχουν χρέη μεγαλύτερα. Οι ίδιες εκθέσεις λένε επίσης σε μας ότι το έλλειμμα σε ένα κύκλο διαρκώς εξελίσσεται και αυξάνεται. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με το έλλειμμα κάτω από 3% και το χρέος λέει που μειώνονται με, μπροστά, αυτά τα στοιχεία, μπροστά σε αυτά τα στοιχεία πρέπει να διαρωτηθούμε. Τι είναι εκείνο που φταίει και δεν αυξάνεται η οικονομία μας. Βρισκόμαστε σε μια λέει τροχιά ανάκαμψης της οικονομίας. Το αντίθετο συμβαίνει. Οι αριθμοί δείχνουν ότι βρισκόμαστε στη συνέχεια του, τέλματος. Και μήπως δεν θα έπρεπε να γίνει μια, ένας αναστοχασμός εκ των υστέρων σύμφωνα με όλα αυτά η λιτότητα είναι εκείνη η οποία περιορίζει και συρρυκνώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να δικαιολογείται ότι πρέπει να εξετάσουμε με σοβαρότητα τον τρόπο να ελαστικοποιήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν είναι οι δυνατότητες δημόσιας, ε, δημόσιων δαπανών, δημόσιων δαπανών για να δημιουργηθούν οι δυνατότητες ε, κρατικής ανάπτυξης ώστε να βρισκόμαστε και εκτός του υπολογισμού της, ε, του ελλείμματος. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διανοιχτεί μέσα από τη συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτό το Ταμείο ε, Επενδύσεων. Η ερώτηση είναι σαφής. Μια και εξακολουθούν και υπάρχουν αυτές οι ανισορροπίες. Αντί να επιμένουμε στην ε, ε, μηχανική, την χρηματοοικονομική μηχανική, θα πρέπει να δούμε μια άλλη εναλλακτική πορεία. Και ουσιαστικά ολοκληρώνω με αυτή την ιδέα θα έπρεπε να ε, ε, δώσουμε προνομιακό χαρακτήρα στις δημόσιες δαπάνες. Να γίνουν έτσι αυτές οι επενδύσεις ώστε να έχουμε με εθνικό στόχο, με εθνικούς στόχους την προοπτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και ο κύριος ε, Βιέγκας εξέφρασε τη διαφωνία του. Επιβεβαιώνω ότι διαφωνούμε ως Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά δεν είναι προσωπική άποψη. Εγώ τηρώ τους κανόνες του συμφώνου και αυτό μου επιτρέπει να μειώσω κάποιες από τις ανισορροπίες και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η καταπολέμηση του δημοσίου χρέους ε, και του ελλείμματος ε, θα έπρεπε να είναι κοινή για όλους ανεξάρτητα με τις ε, πολιτικές μας πεπιθήσεις. Έχουμε χώρες οι οποίες αποδυναμώνονται, υπερχρεώνονται και επομένω επαναλαμβάνω όπως είπα και εδώ αρκετές φορές ότι εάν χρησιμοποιούμε την ευελιξία, είναι στα πλαίσια των κανόνων δεν ε, προσπαθούμε να κάνουμε δημιουργική υπερβολική χρήση της ευελιξίας, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο συμφωνούμε νομίζω, είναι το θέμα των επενδύσεων και νομίζω ότι αυτό αποτέλεσε και κίνητρο του σχεδίου που παρουσίασε ο Ζαν Κλοντιούν και την προηγούμενη εβδομάδα, το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, ε, εφόσον κάποιες χώρες αποφασίσουν να συνεισφέρουν ε, στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων, Αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς του ελλείμματος και του χρέους τους. Thank you. Now for the green, Mr. Ernest Urtasun. Ευχαριστώ κύριος Έρνες Ούρτασομ για τους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη διαδικασία ελλείμματος της Ισπανίας. Το αίτημα σας να μειωθεί το έλλειμμα κατά τέσσερις μονάδες ε, δημιούργησε φυσικά συναγερμό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ευθύνε της Ισπανίας ε, για την κατάσταση του προπολογισμού, υπάρχει και τέλο πάντων είναι δεδομένο. Το να υπάρχει όμως επιπλέον μείωση του ελλείμματος ε, δεδομένη της πολύ σοβαρής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ισπανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι 750.000 νοικοκυριά στην Ισπανία είναι χωρίς κανένα εισόδημα. Είμαστε ε, σε 50% ανέργων που δεν λαμβάνουν κανένα ε, επίδομα. Και επομένω θα πρέπει να γίνει κάτι για να καταπολεμήσουμε την ανεργία και το, ο προπολογισμό τη πολιτική αποσχόληση τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 34%. Η ερώτησή μου είναι, η ε, αίτηση για να μειωθεί το έλλειμμα κατά 0,4% ανέλησε τις κοινωνικές συνθήκες, αναλύσατε τις συνέπειες που θα υπάρχουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας το ποσοστό ανάπτυξης για το τρίμηνο ήταν χαμηλότερο. Είμαστε σε κατάσταση επιβράδυνσης, επομένως αναλύσατε τις συνέπειες ε, ε, του θέματος αυτό, διότι όπως είπατε πολύ καλά κύριε Πίτροπε, υπάρχει μια σχετική ευελιξία που θα μπορούσαμε να την εφαρμόσετε, δεν είναι ανάγκη να εφαρμόζετε κάτι τέτοιο, θα ήθελα να απαντήσετε στην ερώτησή μου και θα ήθελα να ξέρω και την άποψή σας για την ε, δημοσιονομική μεταρρύθμιση της ισπανική κυβέρνησης, η οποία θα μειώσει τα εισοδήματα κατά 9 δισεκατομμύρια θεωρείτε ότι είναι κατάλληλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις ή όχι. Και τέλος, για να ολοκληρώσουμε, όσον αφορά το σχέδιο Juncker, έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι οι εισφορές των κρατών μελών δεν θα ληφθούν υπόψη ή θα υπάρχει κάποια ευελιξία ε, στην ε, υπολογισμό του ελλείμματος. Είναι συνεισφορά σε κεφάλαιο ή μπορεί να είναι και η συνεισφορά ε, σε αγορά ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι αυτό δεν ήταν σαφές στην ανακοίνωση και θα ήθελα να μου το ε, διευκρινίσετε. Λοιπόν, καταρχά, όσον αφορά τον ε, Ισπανικό προπολογισμό, η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών ε, για τι οποίε ε, επισημάναμε ότι υπάρχει κίνδυνο μη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και γνωρίζετε βεβαίω ότι και η Ισπανία έχει μία προθεσμία για να διορθώσει το έλλειμμά τη μέχρι το 2016. Για το 2014 το έλλειμμα θεωρούμε ότι θα είναι κάτω του 5,8% του ΑΕΠ που ήταν ο στόχος. Για το 2015 θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ε, του 4,8 του ΑΕΠ που περιλαμβάνεται στο σχέδιο προπολογισμού της Ισπανίας. Υπάρχει μια διαφορά στους υπολογισμούς μας που οδηγεί σε αυτό το 4,6%. Ε, και εμεί θα συνεχίσουμε να το συζητούμε το θέμα αυτό και να το ζητάμε, διότι θεωρούμε ότι δεν επαρκούν οι προσπάθειες. Υπάρχουν συγκεκριμένε διαρθρωτικές συστάσει. Ε, η Ισπανία γνωρίζω ότι προβλέπει μία μείωση ε, της, ε, του προπολογισμού για την εργασία, που σημαίνει ότι θα έχει συνέπειε στην απασχόληση αυτό και στο κόστος της εργασίας. Και προ αυτή την κατάσταση κατεύθυνση θα συνεχίσει ο διάλογο με την Ισπανία για να δούμε ποια είναι η φύση τη διαφορά που υπάρχει και να ληφθούν ε, ενδεχομένως επιπλέον μέτρα που μπορεί να έχουν ε, και κάποιες συνέπειες και να ε, ακολουθηθούν οι συστάσεις μας που επαναλαμβάνω είναι για να τηρηθεί το έλλειμμα το 2016 και την υπάρχει προσαρμογή. Μιλάμε με τις Ισπανικές αρχές και δεν ένιωσα ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ε, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ ημών και της ε, ε, Ισπανικής κυβέρνησης και δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια στο μέλλον. Ε, τώρα όσον αφορά τις άλλες ερωτήσεις που θέτετε, εξ όσων γνωρίζω ναι, πρόκειται για κεφάλαιο για τις επενδύσεις, αλλά θα πρέπει, δεν ξέρω, έχω ένα επιπλέον λεπτό, θα ήθελα να ξέρω κάτι, διότι δεν μου απαντήσατε, ο κύριο Σουρτασούν, για τη ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Διότι στο σχέδιο προπολογισμού που παρουσιάσατε υπάρχει μια μικρή παραπομπή, καταλαβαίνω ότι είστε απόλυτα ενημερωμένο. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η Ισπανική ε, ε, κυβέρνηση. Κάνει μια ρύθμιση που θα μεταφράζεται σε νέα δις θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε τα πράγματα με βάση και το πνεύμα υπό το οποίο εργαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι για να κρατάει το χεράκι των κυβερνήσεων. Εμεί θέλουμε να γίνονται σεβαστέοι συγκεκριμένοι κοινοί κανόνε και από εκεί και πέρα επαφείται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν τα μέσα για να επιτύχουν του στόχου. Και με αυτό, αυτό το πνεύμα συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν θα ε, κρίνω το συγκεκριμένο μέτρο ή οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Τώρα, ο Μάρκο Βάλλη από το EFTD. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. δημιουργούνται πολύ μεγάλες επικρίσεις για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ε, υπολογισμό του δυνητικού ΑΕΠ και του κενού στο έλλειμμα, ε, που είναι δείκτες για να υπολογίσουμε τον προϋπολογισμό των κρατών μελών. Ο υπολογισμός αυτού του κενού λοιπόν είναι πολύ σημαντικός για να καθορίσει και το ε, πρόγραμμα των κρατών μελών. Και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές αβεβαιότητες σε μια περίοδο οικονομικής αστάθειας όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και ε, η εκτίμηση του Output Gap από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανεξετάστηκε τρει φορέ η εκτίμηση του Output Gap τη Ιταλία για το 2010 και το 2013. Επίση, είναι τελείω διαφορετικό μεταξύ των διεθνών οργανισμών ε, ο υπολογισμό αυτό. Ενώ πέρσι εκτιμούσαμε output cap ε, το 2014 για την Ιταλία μείον 3,6%, όσα υπολόγιζε 0,5,1%. Μήπω θεωρείτε ότι η μέθοδος αυτή είναι παροχημένη και μάλιστα στη στιγμή που το χρειαζόμαστε ε, πάρα πολύ και θεωρείτε ότι η μεθοδολογία αυτή θα μπορούσε να στρεβλώσει σε μεγάλο βαθμό τους υπολογισμούς των ε, προπολογισμών των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα... Όπως είπα πρέπει να είναι σαφής η μεθοδολογία για να προάγει του στόχου που θέλουμε να προαχθούν ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα στο μέλλον. Για την Ιταλία τώρα, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το θέμα που αναφέρατε. Εμείς πιστεύουμε ότι το ΑΕΠ πολιτική γενικά δημοσιονομικά της Ιταλίας ε, ρισκάρει να μην συμμορφώνεται με τις ε, κατευθύνσεις αυτές. Καλωσορίζουμε τα μέτρα ώστε να έχουμε το 3% του ΑΕΠΑ και να μειωθεί το ε, έλλειμμα σε 2,5% του ΑΕΠΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έχει διαθεωτική βελτίωση έναντι του 2014 μέσα στο σημερινό πλαίσιο που γνωρίζουμε με την, ε, το χαμηλό πληθωρισμό και την αδύναμη ανάπτυξη. Έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η, η Ιταλία και το ότι βρίσκεται σε ύφεση η χώρα αυτή επί ολόκληρη σειρά ετών. Τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη και έχουμε συζητήσει με την Ιταλία την δυνατότητα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μείωσης της ανάπτυξης ε, διότι αυτό, θα, ε, αυτό οδηγεί σε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις θα έχει ίσως ένα υψηλότερο έλλειμμα από το 2,7% και μια πολύ μικρή βελτίωση διαρθρωτική στο 0,1% και η δημοσιονομική ε, πολιτική βρίσκεται κάτω από εκείνο το οποίο απαιτείται για να σημειωθεί πρόοδος και είναι ακόμα πιο κάτω από την benchmark της βέλτισες προδιαγραφές για τη μείωση του χρέους σε μια μεταβατική περίοδο. Αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι, θέτουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προκλήσεις στην Ιταλία. Μέσα σε ένα επικοδομητικό πνεύμα συζητούμε την κατάσταση με την Ιταλία και θα συζητήσουμε την κατάσταση ξανά το Μάρτιο 2015 παρακολουθώντας δημοσιονομικά τις εξελίξεις και το πώς προχωρεί το πρόγραμμα. Αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα. Όμως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά, αυτές τις δυσκολίες δηλαδή. Uh, Ευχαριστούμε για το σημείο που αναφέρατε το διαρθρωτικό έλαμα, έλλειμμα. Ο νέος πρόεδρος της ΕΣΓΑΠΑ ε, έκανε εχθές σχόλια που κατευθύνονται προς τη δική σας κατεύθυνση και τα όσα μας είπατε εσείς και ανέλησε πολύ προσεκτικά το θέμα της ε, τρέχουσας μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του διαθροτικού ελλείμματος και σε σχέση με άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Θα υπάρξει λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτό το ζήτημα ούτως ή άλλως. Αυτό Αυτά μας είχε πει ο κύριος Μάρτι Χέτεμέκη. Και θα πρέπει λοιπόν διαθροτικά να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μπάρμπαρα Κάπερ, επόμενη. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Επίτροπε, τα κράτη-μέλη νωρίτερα στο Συμβούλιο μπορούσαν έχοντας συμμαχίες να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων και προστήμων και έτσι να παρακολύσουν τη λήψη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα με την ενισχυμένη πλειοψηφία αυτό είναι δυσκολότερο. Αυτόματα δηλαδή επιβάλλονται ε, κυρώσεις αν δεν υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία εναντίον τέτοιων μέτρων. Υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εντυπωσιακά καταδείξατε πόσα τέτοια τέτοιες δυνατότητες θα τις χρησιμοποιήσετε, δηλαδή θα δίνονται τρίμηνες ε, περίοδοι για να μπορέσουν ε, χώρες οι οποίες κρίνονται ως προβληματικές, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν ε, διατεθεί νωρίτερα, να μπορέσουν να κατατεθούν και με αυστηρότερο πνεύμα θα μπορούν να ερμηνεύονται οι κανόνες και οι κανονισμοί. Ερώτηση, τι εννοείται με αυστηρότερη ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών, ιδιαίτερα με την επιβολή κυρώσεων και προστήμων όταν θα υπάρχει παραβίαση ή παράβαση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερη ερώτηση για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τις δημοσιονομικές ε, εποπτή, την δημοσιονομική εποπτεία όσον αφορά την ε, επιτήρηση Νομίζω είναι ανεπαρκή τα όσα ε, γίνονται. Υποβάλλει την ε, αξιολόγησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να δικαιολογήσουν την στάση τους στα κράτη-μέλη. Δεν λαμβάνεται παρκώ υπόψη το Κοινοβούλιο. Ερώτησή μου, ποιο ρόλο προβλέπετε στο μέλλον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς. Πείτε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, ε, τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκοπεύει να εργαστεί τους επόμενους μήνες. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επαληθεύσουμε τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποιες ε, παρατάσεις, κάποιες προθεσμίες, σας εξηγήσαμε για ποιο λόγο και ε, σας... λέω ότι όλα αυτά θα γίνουν εις βάθος, χωρίς καμία προκατάληψη και τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ε, με βάση συγκεκριμένα γεγονότα, ελήφθησαν ή όχι ε, το 2014 και αν τηρήθηκαν τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν. Και αν δεν ελήφθησαν μέτρα, τότε θα πρέπει να γίνουν επιπλέον προσαρμογές, όπως επίσης θα διασφαλίσουμε ότι οι διαρθρωτικές προσπάθειες οι οποίες ελήφθησαν επαρκούν για να καλύψουν τους στόχους των διαφόρων χωρών, κυρίως της Γαλλίας και ε, αν είναι πάνω ή κάτω από το 0,5% του ΑΕΠ. Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τη, ε, την κατάσταση, τη δυνατότητα της οικονομίας να αντιδρά καλύτερα και να δημιουργήσει μια πιο σημαντική ανάπτυξη. Διότι αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμα οικονομικά πρέπει να υπάρχει ε, πιθανή ανάπτυξη η οποία να είναι πιο ισχυρή. Και αυτό θα κάνουμε στους επόμενους μήνες. Και με βάση τα αποτελέσματα τα οποία θα λάβουμε για αυτές τις τρεις παραμέτρους και επαναλαμβάνω συγκεκριμένε δράσεις, ε, διορθωτικές προσπάθειες και διορθωτικές μεταρρυθμίσεις θα λάβουμε και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Και επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι οι επιθυμητές ε, αποφάσεις. Θέλουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, καλές συμφωνίες και θέλουμε όλα αυτά ε, να τα δούμε ε, σε συγκεκριμένο χρόνο και αν υπάρξουν κυρώσεις δεν απαγορεύεται τίποτα, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συνεργασία μα στου επόμενου μήνε για την οικονομική διακυβέρνηση, για τη δέσμη των δύο μέτρων, για τη δέσμη των έξι μέτρων, για την κυρία Μπερέση η οποία είναι απόλυτα δραστήρια και κινητοποιημένη επί του θέματο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σα ευχαριστούμε σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ για την οικονομική διακυβέρνηση για την έκθεση. Εστέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Διότι ίσως με κάποια καθυστέρηση, αλλά μου έδωσε μια απάντηση στην ερώτηση που είχα θέσει εβδομάδες ή μήνες πριν. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, Επίτροπε, σας είχα ρωτήσει και αναφερόμουν στην ε, Animal Farm του Orwell. Κάποια ζώα είναι πιο ίσα από άλλα δηλαδή σε σχέση με την Επιτροπή. Και φυσικά το αρνηθήκατε αυτό. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τώρα την απάντηση ότι ναι, είναι κάποια ζώα πιο ίσα από άλλα. Και στην κυρία Γκουλάρ απαντώντας λέγοντας ότι ουσιαστικά όλες λέει άλλες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη έβαιναν καλώς εκτός από τη Γαλλία και την Ιταλία. Ε, γι' αυτό χρειαζόντουσαν η Γαλλία και η Ιταλία επιπρόσθετα τρεις μήνες περίοδο. Επιπρόσθετα, έξτρα σοβαρά ουσιαστικά αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι διαφορετικοί κανόνες και κανονισμοί ισχύουν για κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με άλλα. Μήπως εσείς ε, και δίνοντας συνέχεια σε μια ερώτηση που δεν απαντήσατε απόλυτα στον κύριο Φέμπερ για το τι είναι τόσο δύσκολο το 2014 διότι δίνετε αντιφατικά μηνύματα. Αφενός λέτε δεν αλλάζει αυτή η Επιτροπή, δεν κάνει τίποτα άλλο. Κάνουμε λέει τα ίδια όπως και προηγούμενα, η προηγούμενη Επιτροπή. Τώρα λέτε, ναι ακούστε το 2014 ήταν δύσκολο να δοθούν αυτά τα στοιχεία διότι θα αναλάβανε τα ενία νέα Επιτροπή. Μα οι κανόνες και οι κανονισμοί είναι κανόνες και κανονισμοί. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο ποια Επιτροπή είναι στην εξουσία. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι θα είχατε εδώ τα στοιχεία αν, είχε, αν ήταν το 2013 αυτό ή το 2015 και το 2014 ήταν ένα, μια, ένα έτος εξαίρεσης. Γιατί, μα οι κανόνες και οι κανονισμοί είναι σαφείς. Κάνει η Επιτροπή ό,τι κάνει κάθε Επιτροπή. Τι μας λέτε εδώ, είναι πολύ αντιφατικά τα μηνύματά σας. Αυτά ήθελα να πω. Όμως το ότι υπάρχει διαφορά αντιμετώπισης κάποιων κρατών μελών εναντί άλλων κρατών μελών και υπάρχουν κάποια που έχουν περισσότερα δικαιώματα και είναι πιο ίσα από άλλα, θα πρέπει πολύ να μας ανησυχήσει, διότι πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Θέλω να το τονίσω αυτό κύριε. Το υπογραμμίζω. Μπορεί να μην σας αρέσει το ότι εγώ μιλάω ίσια και ξεκάθαρα. Αλλά αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Να δίνονται σαφείς απαντήσεις από την Επιτροπή σε σαφείς ερωτήσεις που ρωτήθηκαν. Και είναι λοιπόν η πολύ ανησυχητική αυτή η απάντηση. Αυτό που θέλω να πω είναι για την ανακοίνωση της επισκόπησης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Τι είπατε εσείς. Είπατε επιλέξει ότι ή πήγαν τα πράγματα καλά ή δεν είχαμε λέει αρκετό χρόνο να τα αξιολογήσουμε τα στοιχεία και κάποιοι κανόνες ε, δεν έχουν λέει δοκιμαστεί μέσα σε κανονικά χρονικά πλαίσια. Αυτά είπατε. Συμφωνώ με, τον, με τα όσα είπε ο Χέρμαν Φαν Δηλαδή ότι η κρίση της, ε, του ευρώ έχει ξεπεραστεί. Αν αυτό σημαίνει ότι επιστρέψαμε σε ομαλή κατάσταση μπορούμε να το συζητήσουμε βέβαια. Είναι όμως ίσως πιο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με την οικονομική διακυβέρνηση υπό ομαλές περιόδους και τι γίνεται σε μια κρίση. Διότι στην κρίση είχαμε αντιπαραθέσεις και διαφορές ε, που δεν έδωσαν την ε, δυνατότητα να είμαστε ενωμένοι. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται υπό ομαλούς όρους και συνθήκες. Και αυτό θα πρέπει ε, χρησιμοποιείται λοιπόν όλο το χρόνο και δεν θα δοθεί απάντηση. Μα ο προηγούμενος αγορητής είχε πέντε λεπτά κύριε. Μα χρησιμο... αν χρησιμοποιήσετε όλο το χρόνο δεν θα υπάρξει χρόνος για απάντηση. Να σας δοθεί απάντηση. Εντάξει θα επιταχύνω λέει ο Μιλήτρια. Για την επισκόπηση αυτή δεν θα πρέπει να είχαμε μια σε βάθος ανάλυση των εξαπλών μέτρων six pack και του two pack ε, των διπλών προτάσεων. Διότι διαφορετικά όλα αυτά είναι βασίζονται στο περιβάλλον εμπιστοσύνης. Αυτά είπε ο Ντράγκη. Και θα πρέπει πραγματικά να τεθούν σε τάξη τα του οίκου κάποιων κρατών μελών. Γιατί διαφορετικά θα υπάρξει νέα κρίση εμπιστοσύνης. Η ερώτηση, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Ποια ελαστικότητα, ποια ελαστικότητα χρησιμοποιήσατε για το παράδειγμα που συζητήσαμε για την Ιταλία και Γαλλία. Κάποιο πρότυπο ελαστικότητας πρέπει να χρησιμοποιήσατε. Ποιο είναι αυτό το πρότυπο ελαστικότητας που χρησιμοποιήσατε. Πιστεύετε ότι περισσότερη ελαστικότητα χρειάζεται ακόμα. Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. 20 δευτερόλεπτα έχετε. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει απάντηση. Κάνατε ολόκληρο λόγο που εκφωνήσατε. Έχω δύο ακόμα ερωτήσεις και δεν φτάνει. Παίρνετε το χρόνο μου πρόεδρε λέει ο Μιλήτρια και δεν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ακούστε λοιπόν. Εντάξει, δέκα λεπτά για την ερώτηση, τρία για την απάντηση. Εσεί λόγο θέλατε να εκφωνήσατε. Ακούσαμε ποιε είναι οι απόψει Τώρα δίνω τον λόγο στον επόμενο αγορητή. Μπορεί να μην σα αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, λέει η ομιλήτρια. ρε, σε επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ. Ίσως μπορείτε να ομαδοποιήσετε για τις απαντήσεις σας, τις παρεμβάσεις αυτές κύριε Μοσκοβισή. Όχι κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω σαφή απάντηση στη δική μου την ερώτηση. Όταν ε, ε, κάναμε τη σχέση μεταξύ τη συζήτηση και την, ε, που κάνουμε τώρα και τη συζήτηση για την ανάπτυξη, μας δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει με πιο ευφυή τρόπο τουλάχιστον το πλωστάσιο που έχετε στη διάθεσή σας και είπατε ότι δεν θέλετε να κάνουμε απλώς μία εξέταση αλλά να έχουμε και κάποια όπλα καθοδήγησης και δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κείμενο το οποίο θα μας παρουσιάσετε, ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν όσον αφορά την ευελιξία, για να διορθώσουμε αυτά τα στοιχεία της οικονομικής διακυβέρνησης, τα οποία ε, είναι ακόμα και σε ε, εμβριακό στάδιο, εμβριακό στάδιο παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσα μέσα στη διάθεσή μας. Όσον αφορά την εφαρμογή σήμερα αυτών των κανόνων, η κυρία Φερέιρα σας ρώτησε για τις ε, διατάξεις των κειμένων που έχουμε ενισχύει και που επιτρέπουν σε έκτακτες περιστάσεις να δοθεί μια περαιτέρω πλοθεσμία στα κράτη-μέλη, αντίθετα με αυτό το οποίο ε, είπαν άλλοι από τους προλαλήσαντες. Όταν παρουσιάσετε αυτό το οποίο θέλατε μέσω της ευελιξίας αναφερθήκατε στις έκτακτες ε, περιστάσεις. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει και μπορούμε να πάμε πιο πέρα και να αποξιολογήσουμε το ρόλο αυτής της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για να δούμε περισσότερο λίγο πράγματα που αφορούν το χώρο, χρονοδιάγραμμα, να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Το είπατε και εσείς ε, στην αρχική σας παρέμβαση αυτό και επίσης να δούμε όπως ε, είπαμε και χθες ε, με τον υποψήφιο και σήμερα πλέον πρόεδρο του ΙΣΕΣΓΑΜΠ, να δούμε τους ορισμούς, ε, είτε για το διαρθρωτικό έλλειμμα, είτε για την ανάπτυξη ε, ή τη δυνητική ανάπτυξη. Ε, το κείμενο το οποίο μας παρουσιάσετε σήμερα όμως για τα δέσμη των 6 συν μέτρων, μας είπε ότι προς το παρόν δεν έχει δοκιμαστεί σε συνήθεις οικονομικές συνθήκες. Μα ακριβώ οι κανόνες αυτοί έγιναν για να αντιμετωπίσουν έκτακτες έντονες περιστάσεις. Επομένως, τι είναι αυτό το οποίο δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε καλά μια κατάσταση που οδηγεί αυτή την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ένα νέο μέσο που είναι το σχέδιο των επενδύσεων. Μας είπατε ότι η αξιολόγηση είναι ε, μία αξιολόγηση ε, προληπτική, εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά σύμμορφη με τη δέσμη των μέτρων και ε, μήπως θα πρέπει να λάβετε υπόψη και τις καλές ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην περιμένετε απλώς την καλή βούληση του, Ευρω... του Συμβουλίου. θα μιλήσω μισό λεπτό για να απαντήσω στην κυρία Ντελάγκε. Νομίζω αν κατάλαβα καλά είναι πέντε λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση. Θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο, επομένως θα μπορέσω να απαντήσω. Ε, όχι, εμείς δεν έχουμε επινοήσει νέους κανόνες και όχι δεν υπάρχει προσέγγιση δύο ταχυτότητων. Ε, το είπαμε και στο Eurogroup και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Δεν θέλω να αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκανε τη δουλειά της και όταν ε, φτάσαμε εμείς σε αυτό το σημείο ο κ. Κατάινεν έλαβε την απόφαση που έπρεπε να, λάλει, να λάβει. Δεν έχουμε ακόμα διαδικασία ε, αυστηρής μη και θα πρέπει να το δούμε αυτό με τις... Ε, κυβερνήσεις που ε, ασχολούνται με το θέμα και θα πρέπει να πω ότι δεν είχαμε ακόμα τα οριστικά στοιχεία και δίνουμε μια προθεσμία ε, μερικών μηνών και αυτό δεν γίνεται για μια προσέγγιση δύο ταχυτήτων αλλά για να δούμε επί ποιας βάσεως θα μπορούσαμε ίσως ενδεχομένως να επιβάλλουμε κυρώσεις. Χρησιμοποιούμε μια τελείως αντικειμενική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτα, απόλυτα διάφανο τρόπο. Δεν έχουμε εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τελείως διαφορετικές ε, πολιτικές ε, ε, προσεγγίσεις, εργαζόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ να πω με την Περβάς Μπερές ότι πρόκειται για κοινή απόφαση. Δεν έχουμε εμεί ορισμό και δεν θα επινοήσω εγώ ορισμό πριν παρουσιαστεί. Πρόκειται για φιλοδοξία ε, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ε, να ε, μη συνειδητοποιούμε και τα όρια που θέσουμε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη και όχι να επινέωσουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα αμφισβητεί τα προηγούμε, το σύμφωνο. Όσον αφορά τις έκτακτες περιστάσεις, ε, να επανέλθω σε αυτό που ρώτησε και η κυρία Φερέιρα. Νομίζω ότι υπάρχουν βελτιώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν και στους υπολογισμούς και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η κάθε κατάσταση και φυσικά και στον ε, τρόπο υπολογισμού του διαρθρωτικού ελλείμματα. Υπάρχουν δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αντίστοιχε και ε, δεν μας δίνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχουν στατιστικά πράγματα αλλά και νεολογικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω και ε, σε περίπτωση ε, στην περίπτωση αυτή μαζί με τον κύριο ε, Ντομπρόφσκης ε, δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει κάποια έκτακτη περίπτωση στην Ευρωζώνη. Τέλος, το τρίτο ερώτημά σας κυρία Μπερές, ε, η κυρία Ντελάνγκη αναφέρθηκε και αυτή ακροθυγό στο ζήτημα, το έχουμε συζητήσει με τον καθένα από εσά, διότι συναντήσαμε και τους δύο. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δύο σταδίων. Ξεκινάμε με ε, τα στοιχεία ε, που έχουμε, την έκθεση που έχουμε τώρα, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε και μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για το μέλλον, η οποία θα περιλαμβάνει και ένα πιο σημαντικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι απόλυτα διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας και με τους υπόλοιπους εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές υπ' αυτό το πνεύμα, ε, αυτό το οποίο μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε η συγκεκριμένη προσέγγιση. Ευχαριστώ, Ντάριος Ροζάτη. Uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Επιτροπέ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση της κυρίας Γκουλάρ και της κυρίας Delange. Θα ήθελα να συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, θεωρώ. Θα πρέπει να αποφύγουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει δύο μετρά και σταθμά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς για τα κριτήρια που χρησιμοποιήσατε για την ε, λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά την παράταση της τελικής αξιολόγησης για τις τρεις χώρες. Αρκεί για ένα μέλος, να μην παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού προκειμένου για να, να πάρει την παράταση αυτή. Ή χρησιμοποιήσατε και άλλα κριτήρια. Θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια προκειμένου να διασκεδαστούν όλες οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες για τη διαδικασία αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Για ένα σημαντικό στοιχείο της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Μία από τις ρήτρε για την, το Σύμφωνο Διακυβέρνησης. Το δημοσιονομικό τμήμα της συνθήκης Μία, ένας από τους όρους εφαρμόζει υποχρέωση στις χώρες να εφαρμόζουν διορθωτικό μηχανισμό στο εθνικό πλαίσιο, το ε, εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να συμμορφούνται με τους δημοσιονομικούς κανόνες και ιδιαίτερα με τον διορθωτικό μηχανισμό σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος. Σας ρωτώ λοιπόν πώς αξιολογείτε τη λειτουργία του μηχανισμού, γιατί έχει εφαρμοστεί από πέρσι ήδη. Πώς αξιολογείται λοιπόν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού και ποιο είναι το καθεστώς εφαρμογής του μηχανισμού σε γενικές γραμμές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο διατυπώσατε την ερώτηση, διότι και πάλι θα είμαι απόλυτα σαφής και πολύ συγκεκριμένος ως προς το τι αποτέλεσε κίνητρο για την, απάντηση, για την απόφασή μας προς αυτή την κατάσταση. Δεν είμαστε στα πλαίσια μιας προθεσμίας, βρισκόμαστε σε μια παράταση η οποία πρέπει να δοθεί για να εξεταστεί με συγκεκριμένο τρόπο ε, η επιρροή τριών παραμέτρων. Το κατά πόσον ελήφθησαν μέτρα για το παρελθόν, για το 2014, για το κατά πόσον η διαρθρωτική προσπάθεια επαρκεί για το 2015 ή όχι και τέλος αν υπάρχουν κάποια διαρθρωτικά στοιχεία, κάποιες παρέμετροι ανάπτυξης που θα πρέπει να τροποποιηθούν για την ε, κάθε χώρα που εξετάσαμε ε, και με την οποία υπήρχε επιπλέον διάλογος ε, εδώ και κάποιους μήνες. Ε, υπάρχει απόλυτη επικοινωνία μεταξύ των δύο επιτροπών και το όσα έκανε ο Γιούρκη Κατάινεν με τον κύριο Μπαρόζο, όλα αυτά ε, τα παρακολούθησε και ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος τότε είχε και καθήκοντα ακόμα και θα αναλάμβανε την Προεδρία. Υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο είναι πιο περίπλοκο για τον κύριο Ντομπρόφσκης και μένα, δεν είναι το κατά πόσον θα πρέπει να καθυστερήσουμε το τάδε σχέδιο προπολογισμού ή το δίνα γιατί υπάρχει ε, πολύ σοβαρή μη συμμόρφωση. Η θέση του κυριου Κατάινεν ήταν σαφής, όχι, κανένας από τους προπολογισμούς δεν πρέπει να παραπευθεί και ε, ε, είμαστε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπρεπε να εργαστούμε από αυτού. Ο Βαλτής Ντομπρόφσκης και εγώ σας διαβεβαιώ για την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα, από το Σεπτέμβριο, γιατί τότε πρέπει να γίνει ο διάλογος προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και για άλλη μια φορά δεν υπάρχει διπλός μηχανισμός, δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν υπάρχει Ευρώπη δύο ταχυτήτων και σας διαβεβαιώ ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν το Μάρτιο θα είναι δεόντως αιτιολογημένες και υπάρχει διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Κανείς δεν αποκλείει να υπάρξουν κυρώσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε πολύ σαφή συμπεράσματα. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλαμε να έχουμε ε, πιο ήπια συμπεριφορά για ε, κάποια χώρα λόγω της θέσης της ε, ή για οποιοδήποτε άλλο. Θέλουμε απλώς να λάβουμε την πιο ευφυή και πιο χρήσιμη απόφαση, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει επιτρέψει να καταλήξουμε στην καλύτερη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, η κύρωση δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις, θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις όταν είναι πολύ σοβαρές οι παραβιάσεις και ε, ε, αμφισβητείται και η αξιοπιστία του συμφώνου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι πάντα είναι καλύτερο να καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα, να έχουμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις και πραγματικές προσπάθειες μέσω διαλόγου και είναι πολύ καλύτερο αυτό από το να έχουμε μια κύρωση η οποία μπορεί να έχει απλό εντελώ αρνητικές συνέπειε. Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, να πω αυτό που είπα και εν γέννη, τα πάντα θα περιλαμβηθούν στην αξιολόγηση που θα κάνουμε για την οικονομική διακυβέρνηση. Είπατε και εσείς ότι πρόκειται για πολύ πρόσφατους ε, μηχανισμούς και αυτή τη στιγμή επιφυλάσσομαι λοιπόν, δεν σας λέω την οριστική ε, κρίση μου επ' αυτού, διότι ε, θα ήταν πρόημο να σας πω οριστική άποψη τώρα. Ευχαριστώ, Ούντα Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ανταλλάξουμε παρατηρήσεις και να θέσω μια ερώτηση. Η παρατήρηση που θέλω να προσφέρω είναι η εξής. Νομίζω η Ευρώπη γνωρίζει δύο ομάδες προβλημάτων. Αφενός ε, ιδεολογικά θέματα, ιδεολόγοι. Είναι εκείνοι οι οποίοι άσχετα ποια οικονομική πραγματικότητα έχουν μπροστά τους, άσχετα αν βρέχει, χιονίζει ή λάμπει ο ήλιος, έχουν ε, την πραγματικότητα που θέλουν να την υποτάξουν στα ιδεολογήματά τους. Πάντα ίδιε ίδιες δίνονται. Περικοπές λέει δημοσιονομικές, άσχετα ποια είναι η οικονομική βάση. Έχουμε τέτοιους ιδεολόγους στη χώρα μου. Κάποιοι άλλοι υπάρχουν σε άλλες χώρες. Υπάρχουν και στη γενική σας διεύθυνση τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν άλλοι που δεν ζήτησαν καν συγγνώμη για όσα συνέβησαν με την Τρόικα στην Πορτογαλία και άλλες χώρες, όπου υπέστησαν πλήγματα, όπου διαγράφηκαν, εξαλείφθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις. Αυτή είναι η ιδεολόγη. Δεύτερη ομάδα είναι εκείνοι που αρνούνται τον εξυγχρονισμό. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν τίποτα καινούριο. Θέλουν να συνεχίσουν με αυτά που έκαναν. Ζούνε σε μια ενιαία αγορά, λέει, με 28 κράτη-μέλη. Αδιάφορο λοιπόν να αφήσουμε τα πράγματα όσοι είχαν. Αυτό πιστεύω ότι αυτό θέλω να συνεισφέρω στη συζήτηση, αυτό να εισαχθεί. Να δούμε την αντιστοιχία αυτών των δύο προβληματικών ομάδων. Με, αυτή, με σε αυτό το πεδίο έντασης αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη ή η αεριοσπαστική δεξιά. Πρέπει να διαρρήξουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Τίθεται το ερώτημα. Γιατί με τη βοήθεια των υπηρεσιών σας δεν γυρνάμε στους παλαιούς αξιόπιστους αριθμητικούς υπολογισμούς και μαθηματικούς υπολογισμούς με στοιχεία τα οποία είναι αξιόπιστα και γιατί δεν υποβάλλεται άμεσα μια μελέτη. Ε, και τότε θα μπορούσατε να εξηγήσετε το τι έγινε και τι γίνεται τρεις ε, υπολογισμούς να κάνετε σε τρεις φάσεις ανάπτυξης με τα στοιχεία των οικονομικών στοιχείων που αναμένουμε. Την φάση ανάπτυξης. Κάθε χώρα αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύει ένα συγκεκριμένο ποσοστό περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα και υπολογίζουμε συσσωρευτικά αποτελέσματα να το κάνουμε αυτό. Δεύτερη εξελικτική φάση. Κάθε χώρα θα επενδύει ένα συγκεκριμένο ποσοστό παραπάνω και θα κάνουμε τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Όπως το πρόγραμμα με τον χρονορίζοντα 2020 από κοινού με εμάς σχεδιάσατε και θα υπολογίσουμε συσσωρευτικά και θα κάνουμε μετά το status quo υπολογισμό χωρίς πρόγραμμα Juncker, χωρίς επενδύσεις και πρόσθετα από τα κράτη-μέλη. Και σε αυτές τις τρεις εξελικτικές φάσεις θα κάνετε μια προοπτική για το πώς θα έχει το, κρά... το χρέος σαν κράτη-μέλη και θα ξέρουμε για ποιο πράγμα συζητάμε και θα ξέρουμε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε θεσπιστούν οι κανόνες και οι κανονισμοί και τι θα κάνουμε με τις αρχές και τις ιδεολογίες μας για να μπορέσει επιτέλους να αναπτυχθεί η Ευρώπη και να περάσουμε από τη φάση χρεών σε ένα καλύτερο διάδρομο και καλύτερη οδό ανάπτυξης και απασχόλησης. Θα σας παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε το ανθρώπινο δυναμικό σας, μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνετε αυτές τις αναλύσεις και θα έχουμε μια νέα βάση συζήτησης για του χρόνου. Δεν μπορώ εδώ να εκφράσω πολιτικές ε, ιδεολογικές απόψεις. Εγώ είμαι εδώ για να γίνονται σεβαστή κάποιοι κανόνες. Η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ, ε, στις οποίες έχω την ευθύνη, ε, και υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που έχουν κάνει μακροοικονομικές μελέτες και δέχομαι την πρότασή σας με πολύ ενδιαφέρον. Θα την εξετάσουμε. Ο Αλέλα Μασούρ στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρόσεξα, κύριε Επίτροπε, τις απαντήσεις που δώσατε στις διάφορες ερωτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης ενώπιον κάποιων χωρών. Θα σας πω ένα προσωπικό μου φόβο. Πριν από 11 χρόνια, το σύστημα που τότε αποκαλούσαμε κριτήρια του Μάστριχτ, ε, πολυμερούς εποπτείας και υπορβολικού ελλείμματος απέτυχε παταγωδός διότι η Γερμανία και η Γαλλία παραβίαζαν το σύστημα ταυτόχρονα και βρέθηκε μια πολιτική λύση η οποία όλο τυχαίω επέτρεψε με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία να μην επιβληθούν κυρώσεις σε αυτές τις δύο χώρες. Έκτοτε ενισχύσαμε αφενός την πειθαρχία, τη διαδικασία των κυρώσεων, ε, τέθηκε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το ευρωπαϊκό εξάμεινο και το καθεξής. Αλλά πολύ φοβούμε ότι το πολιτικό εμπόδιο το οποίο αντιμετωπίσαμε πριν από 11 χρόνια θα ξανάρθει αύριο και θα βρεθούμε ενώπιον ενός φαινομένου too big to fail, οι μεγάλοι δεν αποτυγχώνουν, που θα ήταν ε, για τις χώρες too big to be blamed σε αυτή την περίπτωση. Μπορούμε κάλλιστα να κατηγορήσουμε την Ιρλανδία, μπορούμε να, καταλα... Ε, να κατηγορήσουμε ακόμα και την Ισπανία και έρχομαι σε αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Ουρτασούν. Αλλά από την Ιταλία και μετά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούμε πια να τις κατηγορήσουμε και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς σταθερότητας. Και μάλιστα οι τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία δεν θα τιμωρηθούν ποτέ. Ελοχεύει ο κίνδυνος λοιπόν να βρεθεί μια κατάσταση ε, εντός της οποίας στην πραγματικότητα, επειδή φοβόμαστε να ξυπνήσουμε τις αγορές, εάν τα επιτόκια της Ελλάδος ε, ε, και τα spread φτάσουν στο 8% μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά αν ξυπνήσουν οι αγορές για τις μεγάλες χώρες, η Ευρωζώνη θα απειλείται εκ νέου και επομένως ελοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούμε ενώπιον μιας κατάστασης πολύ μεγάλης ανισότητας που σοκάρει μεταξύ αυτών που λόγω της ε, πολιτικής του σημασίας έχουν τη δυνατότητα να μην τιμωρηθούν και αυτών που ε, μεσοπρόθεσμα μπορεί να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία του συστήματος. Ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ, ο κύριος Μουσκοβησή. Θα πρέπει να πω και πάλι ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Εγώ θεωρώ και είμαι πεπισμένος ότι η κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμη με αυτό το οποίο συνέβη ε, στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κάτι ε, τέτοιο και σας εξήγησα ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι που μας οδήγησαν ε, στην παράταση κάποιων μηνών. Σας εξήγησα τι θα συμβεί σε μερικούς μήνες. Θα υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος που θα μας οδηγήσει στις μεταρρυθμίσεις και αυτό επιθυμώ και αν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν είναι σε καμία περίπτωση λογικής ε, to be to be blamed. Το επαναλαμβάνω και πάλι. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να επισημαίνω. Μία πιθανή αντίπαση μεταξύ αυτών που είπατε και αυτό θα ήθελα να το σκεφτείτε. Ε, το να υπάρξουν πιθανέ κυρώσεις και δραματικές συνέπειες για τις αγορές ε, ε, και για την Ευρωζώνη συγκυριακά μας οδηγεί στο κατά πόσον θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Εγώ δεν συμφωνώ με την ε, ε, διάγνωση που κάνετε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις και να δούμε και από εκεί και πέρα σε τι θα μας οδηγήσουν. Και υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Από την αρχή της ε, ακρόασης, αυτό κάτι μου υπενθυμίζει, αναφερόμαστε στην κατάσταση μιας χώρας, την οποία εσείς γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Λαμασούρ, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πιο αυστηροί με τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο από ότι με τους άλλους. Υπάρχουν 7 χώρες, όχι 3, 7 χώρες οι οποίες κινδυνεύουν να μη συμμορφούνται. Και οι 3 χώρες τις οποίες ε, έχουμε δώσει ραντεβού το Μάρτιο, πολύ συγκεκριμένα και το επαναλαμβάνω, χωρίς ε, καμία ε, προκατάληψη, είναι η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Και μάλιστα αυτό είναι το ραντεβού της αλήθειας. Δεν είναι για να είμαστε πιο ήπιοι, πιο διαλλακτικοί, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστία, υπάρχει αξιοπιστία για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αξιοπιστία για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοπιστία για τον Επίτροπο, για του επιτρόπου που είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά, τον υποφαινόμενο, το συνειδητοποιώ απολύτω και επειδή ακριβώ το συνειδητοποιώ απολύτω, ε, σα λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Θα τι αναλάβουμε σίγουρα. Ευχαριστώ, Άλφρετ Σάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αφενός δηλώνουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τη μείωση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να ενισχύσει την δημόσια και την ιδιωτική επένδυση. Και στο μεταξύ ε, το 2 και το 6 στοχεύουν τις, ε, τα υπερβολικά ελλείμματα σε μια κατάσταση όπου δεν βασιζόμαστε στους υπολογισμούς στην ε, πραγματική κατάσταση. Και φυσικά είναι πιο εύκολο για τις κυβερνήσεις να κόψουν τις επενδύσεις ανά παρά να κόψουν τις τρέχουσες δαπάνες. Το 2 και το 6 λοιπόν υποτίθεται ότι θα ε, ενίσχυαν τι επενδύσεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για αυτή την αντίφαση. Δεύτερη ερώτηση για τις συστάσει αναχώρα. Επειδή υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά του προπολογισμού που έχουν παρουσιάσει τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε τα τεχνητικά κριτήρια που θα πρέπει να καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι συστάσει τη. Όταν κάνει όμω εκτιμήσει, πάντα υπάρχει ένα υποκειμενικό παράγοντα. Το ερώτημα παραμείνει λοιπόν. Μιλάμε για την Ευρωζώνη στο σύνολο της εκτιμήσεις ή μιλάμε για την εκάστοτε χώρα. Γιατί μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και τα δύο συνάδουν. Αλλά μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Ποια είναι η ισορροπία μεταξύ των εθνικών συμφερόντων των χωρών και της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Αυτό έχει να κάνει και με την όλη αντίφαση του τι κάνουμε με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά θεωρώ ότι αποτελεί και ένα αυτοτελές ερώτημα. Η απάντηση. Κοιτάξτε, ειλικρινά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της εφαρμογής των κανόνων και του σχεδίου επένδυσης. Όπως είπε και η κυρία Περές πριν από λίγο, όπως αποκοινούμε τους επιτρόπους τα Ισαν και να σας παρουσιάσουμε την ε, μελέτη ετήσιας ανάπτυξης ε, ως ε, μια συνολική προσέγγιση από τρεις παράγοντες. Η δημοσιονομική πειθαρχία, διαστατικές μεταρρυθμίσεις και τρίτο σκέλος είναι το καινούριο σκέλος, το επενδυτικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλα αυτά αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι απόλυτα απαραίτητο να συνεχίσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία. Και επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό ότι το να υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα και να υπάρχουν μεγαλύτερα χρέη δεν είναι το δυνατό σημείο μιας οικονομίας. Κοιτώντας τις δημόσιες δαπάνες για τις επενδύσεις. Το επενδυτικό λοιπόν πρόγραμμα, όπως ξέρετε, σχεδιάστηκε με τη σύσταση ενό ταμείου που βασίζεται σε εγγύησει από το Ευρωπαϊκό προπολογισμό και στην εφαρμογή του κεφαλίου του EIB+. της Ευρωπαϊκής τράπεζες Τράπεζας. Ποσών που δεν θα συμπεριληφθούν στο έλλειμμα ή στο χρέος των χωρών. Αυτή είναι η γενική προσέγγιση. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη γιατί πολύ απλά χρειάζεται πιο μεγάλη συνοχή και γιατί πραγματεύεται όλες τις πτυχές της λύσης που καλούμαστε να βρούμε για να βγούμε από την κρίση. Χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλή ανάπτυξη και υψηλή ανεργία. Απαράδεκτα όλα αυτά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επαναλαμβάνω λοιπόν για το δεύτερο ερώτημά σας ότι μέσω του σχεδίου τη γραμματότησή μα για το σχέδιο προπολογισμού και μέσω τη διαδικασία ανισορροπιών έχουμε αναλύσει την σχετική κατάσταση πιστωτών και χρεωστών και ξέρουμε λοιπόν ότι θα χρειαστούν προσπάθειε και από τι δύο πλευρέ και ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερο συντονισμό τη οικονομική πολιτική και ότι επίση χρειαζόμαστε σε κάποιε χώρε έρευνα της ε, δημοσιονομικής ικανότητας σε ό,τι αφορά και τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Ευχαριστώ όλοι. Ο Πρόεδρος, τελευταίος ομιλητής τώρα, ο Κούναρ Χοκμάρκ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Επίτροπο. Πολύ μεγάλο μέρος της συζήτησης γύριζε γύρω από τις απόψεις ε, για τα ελλείμματα Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν παρεκκλήσεις, αποκλίνουσες απόψεις εδώ. Κάποιοι λένε ότι κάνουμε λόγο για δογματικούς πολιτικούς έναντι άλλων που είναι πραγματιστές. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε την πραγματικότητα. Όταν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επετράπη στη Γερμανία και τη Γαλλία να έχουν ελλείμματα, δημιουργήθηκαν προβλήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι κυβερνήσεις ήταν εκείνες που είχαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα αυξημένα ελλείμματα και μετά δεν είχαν χρήματα πια και άρχισε η περίοδος λιτότητας και περικοπών δεν είχαμε την δυνατότητα να είναι αηφόρος η πολιτική των παγιωμένων ε, προϋπολογισμών και δημοσιονομικών. Είχαμε ε, οικονομίες ε, που είχαν αποτελματωθεί και δημιουργήθηκε ύφεση. Βλέπουμε την άνοδο των εξτρεμιστών. Βλέπουμε ότι στις χώρες που έχουν αυξημένα ελλείμματα ότι υπάρχουν ακραίες τέτοιες τάσεις. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί αυτό αφορά την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τι κάνετε με τα ελλείμματα. Διότι ε, συζητούν κάποιοι και λένε εντάξει ας υπάρξουν ελλείμματα με την ελπίδα ότι θα δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη έχουν όμως αρνητικά, ε, αρνητικές επιπτώσεις τα ελλείμματα. Οι χώρες με τα, με τα περισσότερα ελλείμματα είχαν ε, την ε, ανάπτυξη και την δυνατότητα προοπτικής θετικής. Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα των ελλημάτων. Ο λόγος να υπάρχει ένα σύστημα σταθερότητας, ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης να ελέγχονται, είναι να ελέγχονται τα αρνητικά εκείνα φαινόμενα που υπονομεύουν το πνεύμα του επιχειρήν, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τι πιστεύετε εσείς, πώς το βλέπετε και αναλύετε το θέμα των ε, ελλημάτων εσείς. Ελπίζετε ότι με την ε, αναβολή πολιτικών για να μειωθούν τα ελλείμματα μπορεί να βοηθήσει χώρες να έχουν ανάπτυξη κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν να κερδίσουν και να πετύχουν επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ή βλέπετε τα ελλείμματα ως πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτως ή άλλως επιτέλους. Και τελευταία ερώτηση, αν δεν υπάρχουν πρόστιμα και κυρώσεις για αυτή την παρατεταμένη περίοδο που υπήρχαν ελλείμματα και ήταν τόσο παρατεταμένη, τα είδαμε τα ελλείμματα επί μεγάλη περίοδο χωρίς καμία αντίδραση από πλευρά σας. Δηλαδή η μη επιβολή κυρώσεων και προστήμων μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας ή όχι. Πώς το βλέπετε. Διότι η αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας είναι κάτι το οποίο μας βοηθά όλους. Μπορεί να μας βοηθήσει, είναι κέρια σημασίας για την δυνατότητα δανειοληψίας, ε, πιστώσεων για την ανάπτυξη. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα της αξιοπιστίας. Με αυτή την ευκαιρία θα να επαναλάβω ένα μήνυμα το οποίο είχε γίνει ούτως ή άλλως κατά την έναρξη αυτής της συζήτησης και προηγούμενα. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή δεν μπορεί να έχει δόγματα. Λειτουργεί με βάση εφαρμογή κανόνων και κανονισμών, με ένα πραγματιστικό πλαίσιο και νοοτροπία. Να είναι απόλυτα σαφές αυτό. Είμαι απόλυτα δεσμευμένος για την μείωση των ελλημάτων και των χρεών. Πιστεύω ότι το χρέος και τα ελλείμματα δεν είναι λύσεις για μια ανταγωνιστική οικονομία χρέη και ελλείμματα είναι εχθροί της οικονομίας και της ανάπτυξης. Και όταν υπάρχει μεγαλύτερο χρέος και έλλειμμα, τότε μια οικονομία αποδυναμώνεται. Δηλαδή, πόροι για την εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους είναι κάτι που χάνεται και δεν μπορεί να δοθεί στην ανάπτυξη. Ξέρω ότι κάποιες χώρες ε, με τα ελλείμματα αυτά ε, θα πρέπει να μπορέσουν να οδηγηθούν σε καλύτερα αποτελέσματα από μας. Δεν είμαστε σε μια διαδικασία παράτασης ή αναβολής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τρεις μήνες δόθηκαν όλοι για να εξεταστεί σε βάθος ακριβώς η κατάσταση τριών χωρών όλων και όλων. Και αυτό θα το κάνουμε χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε χαλαρότητα ή ε, αυταρέσκεια. Αυτό ήθελα να πω και θα δώσω και την τελική μου παρατήρηση τώρα. Προσωπική μου πεποίθηση είναι και θα δώσω αγώνα να εφαρμοστεί αυτό. Ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις και να γίνουν ε, δράσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ε, αντιμετωπίζοντας χρέη και λύματα. Αν μπορούμε να αποφύγουμε κυρώσεις και πρόστιμα πετυχαίνοντας αυτόν τον στόχο πάντα είναι καλύτερο, χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις. Αν όμως θα είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα επειδή ο διάλογος δεν οδήγησε σε χειροπιαστά αποτελέσματα και στα αναμενόμενα αποτελέσματα, ε, τότε λοιπόν θα υπομισθούμε την ευθύνη και θα επιβάλλουμε κυρώσεις και πρόστιμα. Αυτή είναι η προσέγγιση την οποία υιοθετούμε και ο Βάλτης Νταμπρόφσκης και, και, και εγώ μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεών μας. Να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα αποτελέσματα των διαλόγων μέχρι σήμερα εξετάζοντας τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια αν αυτοί οι διάλογοι είχαν τελεσίδικα αποτελέσματα, καθοριστικά αποτελέσματα, τότε δεν θα δίναμε περισσότερο χρόνο για να εξετάσουμε κάτι. Αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι έπρεπε να επιβληθούν προ, ε, προς, προς πρόστιμα και κυρώσεις θα το είχαμε κάνει. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η αμφιβολία ε, λάβαμε την απόφαση να δοθεί μια μεταβατική περίοδο σε ένα διάστημα μικρό για να τα ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε Μοσκοβισή, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωντανή και χρήσιμη συζήτηση αυτός ο διάλογος. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει πιο μπρος από τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να βρεθεί κοινό έδαφος για την υλοποίηση μιας νέας στρατηγικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να εργαστούμε και εμείς και να προσπαθήσουμε με βάση αυτό το διάλογο να συναγάγουμε συμπεράσματα και για τη δική μας δουλειά και με βάση κάποια γεγονότα τα αντικειμενικά στοιχεία που πρέπει να θυμόμαστε. Το πρώτο, το ότι δεν είμαστε στην νομική κατάσταση του 2003 και αυτό χάρη σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Και για την έκθεση Βόρτμαν Call που εισήγαγε σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το άρθρο 5 που ζητεί να λαμβάνεται υπόψη ότι κάποιες εξαιρετικές ε, κατεξαίρεση καταστάσεις και μ, μεταρρυθμίσει ε, που έπρεπε να γίνουν και οι προηγούμενοι δεν είχαν καθορίσει με ποιες διαδικασίες ε, οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υπολογίζονται και αν μπορούν να επιτρέψουν να υπάρξει ένα μεσοδιάστημα για να γίνει κάτι. Αυτή είναι η δουλειά λοιπόν η δική μας και της νέας επιτροπής. Σε αυτό το μη ολοκληρωμένο έργο, αν το έργο, να δώσουμε συνέχεια να ολοκληρωθεί. Αυτή η διάταξη δεν υπήρχε το 2003. Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε λοιπόν με διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικά πράγματα. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι 7 χώρες 7 χώρες εξετάστηκαν ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της μη συμμόρφωσης και τρεις επελέγησαν ως εκείνες που βρίσκονται εν δυνάμει ενώπιον νέων λήψης νέων μέτρων ή νέ, ε, ε, κάποιων μέτρων και δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι υπήρξε ξεχωριστή αντιμετώπιση αυτών των τριών έναντι των άλλων τεσσάρων που ε, είχε αρχίσει μια νέα φάση ε, ειδική επιτήρησης. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια νέα φάση πραγμάτων. Αυτό να το λάβουμε υπόψη και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και με βάση τη νέα μακροοικονομική στρατηγική που σαφώς καταδείχθηκε και εξετάστηκε, παρουσιάστηκε από τους τρεις επιτρόπους, θα προχωρήσουμε προχωρήσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Μοσκοβισή, του συναδέφους. Προχωράμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξη. Σα ευχαριστούμε κύριε Μοσκοβισή. Για το τελευταίο αυτό σημείο πρέπει να ζητήσω συγγνώμη αλλά και να παραπονεθώ σε σχέση με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου διότι προφανώς δεν ήταν σε θέση το Κοινοβούλιο να παράσει διερμηνία για την τελευταία ώρα α, των δραστηριοτήτων αυτής της Επιτροπής και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέχρι τις 12.30 θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε τώρα για την ε, μηνιαία επισκόπηση των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων που είναι πολύ σημαντική υπόθεση για τις δραστηριότητές μας. Τελειώσαμε εδώ έτσι. Και ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις είναι κέρια σημασίας και σε σχέση με το επίπεδο παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα αρνητικό το ότι οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου δεν παρήχαν, δεν παρέσχαν ε, δυνατότητε διαρμηνία ε, για αυτή μα τη συνεδρίαση, για αυτό το θέμα. Παραπονούμαστε, πρέπει να εκφράσουμε το παράπονό μας από κοινού. Και τερματίζουν εδώ οι διερμηνείς, ευχαριστούμε.